ξεκινάμε εκ νέου τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα εγκεκριμένα κείμενα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν παρατηρήσεις. Έχετε παρατηρήσεις? Όχι, εντάξει. Τα πρακτικά εγκρίνονται. Τώρα περνάμε στο πρώτο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης, της απογευματινής, που είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. εκπροσωπηθεί η ύπατη εκπρόσωπος από τον Επίτροπο Γιώχανες Χάν που έχει και το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας και θα πρέπει να τα σεβόμαστε και να διώκουμε τις ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αποτελεί μέρος της καθημερινής εργαλειοθήκης και θα πρέπει και οι εταίροι μας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Αυτή η εργαλειοθήκη είναι συνεκτική και λαμβάνει υπόψη την πολύ πλευρή και διμερή διάσταση. Θα καταδικάζουμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και να λαμβάνει η χώρα και θα θέλαμε να υπάρχει λογοδοσία των χωρών. Φυσικά η παγκόσμια σκακέρα εξελίσσεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό ε, έχουμε προβάλει μία στοχοθετημένη αποτίμηση που θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία στις συλλογικές προσπάθειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, δίωξη των παραβιάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το μελλοντικό καθεστώς για να δούμε ποιες παραβιάσεις εμπίπτουν σε αυτό το καθεστώς. Εκεί που υπάρχει συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκεί που υπάρχει διαφθορά και παραβίαση του ανθρωπίνου δικαίου, εκεί θα πρέπει να υπάρχει μία διάδραση και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τα Ηνωμένα Έθνη. Οι παραβιάσεις ε, λαμβάνουν υπόψη την ε, γεωγραφική διάσταση Μιανμάρ, Ιράν και Δημοκρατία του Κονγκό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν ε, βεβαίως χάσματα γιατί η γεωγραφική διάσταση είναι περιορισμένη θα μπορούσαμε να έχουμε ένα οριζόντιο καθεστώς ε, ε, δίωξης των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχουμε μια εύρωστη πολιτική για να γίνουν και προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το ΕΔΑΔ. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις σφαιρικές αρχές που ισχύουν για την κύρωση των παραβιάσεων μέσα στα πλαίσια του δικαίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι γιατί γίνονται συζητήσεις εμπειρογνωμόνων για να διευκρινίσουν όλα αυτά τα θέματα. Τη στιγμή που θα δοθεί τελική μορφή στη συζήτηση θα γίνουν συζητήσεις πολιτικής υφής. Τα 28 κρατη θα πρέπει να συμφωνήσουν ομοφόνος για αυτό το καθεστώς, όπως ισχύει για συγκεκριμένες κυρώσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας και προσβλέπω στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα η κυρία Καλινέτε Σάντρα να λάβει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, μερικές φορές ε, ένα όνομα σημαίνει πάρα πολλά. Ε, ονομάσει κανείς ε, το καθεστώς αυτό με βάση τον κύριο Μαγνίτσκι, αυτό θα ήταν ένα αμφίσιμο μήνυμα. Ε, θα μπορούσε να προκληθεί εντύπωση ότι η Ευρώπη ε, θα προκαλέσει πολλές και σοβαρές συνέπειες για εκείνους αλλά και για πολλούς άλλους στον κόσμο. Ο Μαγνίτσκι στάθηκε κατά του καθεστώτος Πούτιν. Ο τρόπος με τον οποίο η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει την δολοφονία του, αυτό κατέστη το σύμβολο της ατιμορρησίας. Γι' αυτό λοιπόν Λοιπόν, το όνομα του Μαγνίτσκι ε, είναι σημαντικό για όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι το ότι καλούμε το να υπάρξει ένα, μια ευρωπαϊκή πράξη Μαγνίσκη. Αυτό σημαίνει νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων ε, και για το πάγωμα των ε, τραπεζικών λογαριασμών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρχει ε, τιμωρησία για δολοφόνους πουθενά, ούτε και στην Μιανμάρ, αλλά ούτε και στην Κεντρική Αφρική ή στους δολοφόνους των δημοσιογράφων. Για άλλη μια φορά θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση για να υπάρξει πράξη Μαγνίσκη πριν από το τέλος της θητείας. Μέχρι τώρα το Συμβούλιο δεν δραστηριοποιήθηκε, αλλά τώρα αυτή η πρωτοβουλία κερδίζει περισσότερο σε ενθουσιασμό. Η κυρία Γκόμες... Το Κοινοβούλιο το 2013 στυλίτευσε τη διαφθορά στις τρίτες χώρες. Ήμουν εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να, εγκρίνει, όπως έκανε και η ΕΠΑ, την λεγόμενη πράξη Μαγνίτσκι περί λογοδοσίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ασχολήθηκε με το θέμα λογοδοσίας ως προς την δολοφονία του Σεργέη Μαγνίτσκι και τη λογοδοσία γενικότερα τρίτων χωρών για να γίνονται, να δακτυλοδεικτούνται μάλλον οι παραβιάσεις και η διαφθορά. Έξι χρόνια μετά έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό. Μιλάμε για την πράξη Μαγνίτσκι, γιατί αυτή η δολοφονία έγινε στη Ρωσία του Πούτιν αλλά θα μπορούσε να ισχύσει οπουδήποτε. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις, γιατί δυστυχώς πολλές χώρες είναι όμοιροι, πολλές χώρες είναι όμοιροι ολιγαρχικών καθεστώτων που είναι ουραγή του Τραμπ. Μην ξεχνάμε την ε, δολοφονία της δημοσιογράφου από τη Μάλτα, καθώς και άλλες δολοφονίες ε, δημοσιογράφων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπασίρ για ένα λεπτό. Chair, Commissioner Milton Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαν, ο Μίλτον Φρίντμαν έλεγε ότι ένα μεγάλο λάθο είναι να κρίνουμε τι πολιτικέ και τα προγράμματα από τι προθέσει του και όχι από τα αποτελέσματά του. Από την αρχαία Ελλάδα και του πολυπονησιακού πολέμου έω τη Λευκορωσία, το Ιράν και τη Μιαμάρ και τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία σήμερα, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι οι κυρώσει απέναντι σε χώρε ολόκληρε σπάνια πετυχαίνουν τους στόχους εξωτερικής πολιτικής. Πολύ συχνά οι συλλογικές αυτές τιμωρίες οδηγούν σε μεγαλύτερη συσπήρωση και οι αθώοι πολίτες σε αυτές τις χώρες εξαρτώνται ακόμα περισσότερο από τους δυνάστες του σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε βασικά αγαθά. και βεβαίω έτσι περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι πολιτικέ και κοινωνικέ του ελευθερίε. Εγώ ω υπέρμαχο τη ελεύθερη αγορά ήμουν πάντα υπέρ τη ατομική ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα, μια έξυπνη πολιτική κυρώσεων για να εξασφαλίσουμε ότι οι κυρώσει αυτέ θα είναι στεναρέ, αλλά και αποτελεσματικέ απέναντι σε όσου έχουν προβεί σε καταχρήσει ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπασίρ. Η κυρία Σάκε έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανεί ότι έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε που έχω υποβάλει τροπολογίε ε, για την, ε, ε το νόμο Μαγνίτσκι. Θέλουμε έναν έξυπνο μηχανισμό έτσι ώστε όσοι παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα ατομικά να μπορούν να λογοδοτήσουν. Αυτό επήγει ακόμα περισσότερο σήμερα από ό,τι τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Τομέων Εθνών και τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα συχνά παραλύουν λόγω των βέτο που υπάρχουν, πρέπει να μπούμε στην πρώτη γραμμή και να μπούμε σε αυτή τον ασπισμό των πρόθυμων. Οι Ηνωμένες Καναδά, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες της Βαλτική ήδη έχουν νομοθεσίε τύπου Μαγνίτσκι. Εστιασμένες ε, ε, κυρώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με πάγωμα λογαριασμών, απαγόρευση εισόδου, ε, για αυτούς που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, είτε είναι κρατικοί φορείς είτε όχι, μπορεί να, κάνουν μεγάλη, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και για να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ της τιμωρία ατόμων από το να ε, τιμωρούνται ολόκληροι λαοί. Οι ελίτ είναι αυτέ που συχνά συμμετέχουν σε αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στέλνουν συνήθω τα παιδιά του ε, στα καλύτερα, καλύτερα πανεπιστήμια τη Ευρώπη και έρχονται για ψώνια εδώ. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτό για ανθρώπου που έχουν δολοφονήσει ε, δημοσιογράφου ή έχουν βιάσει γυναίκε. Όταν μιλάμε λοιπόν για καθεστώ κυρώσεων, πρέπει να εξετάσουμε και εμεί τον εαυτό μα. Έτσι, διότι πέρα από τι κυρώσει που υπάρχουν, υπάρχουν εταιρείε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργούν γέφυρες ε, στο Κούρσκ, στα στενά του Κούρσκ, άλλοι συνεργάζονται στη Συρία με τρομοκράτε. Δεν, μπορούμε λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι, δεν μπορούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι από τον πιο αδύναμο κρίκο στι συμπεριφορέ μα. Τελειώνοντα, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα οριζόντιο σύστημα κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά το πιο βασικό είναι να μπορούν να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν τα εγκλήματα αυτά σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια. Πρέπει να σταματήσει η ατιμορρησία και εγκρίνοντα το κανονισμό αυτό θα έχουμε κάνει και εμείς ένα μικρό βήμα για τη δικαιοσύνη και για τη Σάρβεϊ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόχμπιλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε με το να υπάρξει ένας ε, μηχανισμός ε, που θα τιμωρεί τους υπεύθυνου. Αν το κάνουμε αυτό θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει πάντα να διώκονται. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ποινική δίωξη των δραστών αλλά θα πρέπει να υπάρξει δίωξη ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι δράστες κατορθώνουν να ξεφύγουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εδώ και καιρό εφαρμόζει βάζει ε, συγκεκριμένες κυρώσεις ε, κατά προσώπων. Αυτό έγινε την πρώτη φορά όταν ε, όταν κρεμάστηκε ο Νιγηριανός ακτιβιστής το 1995. Σήμερα λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι να απαγορεύουμε την είσοδο και να παγώνουμε τους λογαριασμούς των δραστών και αυτό να γίνεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σωστό το ότι θα μπορούν και να ε, να εφεσιβάλλονται οι κυρώσεις, αυτά βέβαια ε, να, γίνονται, να δημοσιοποιούνται στην κοινή γνώμη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα εάν δεχτούμε και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Κυρία Λόχμπιλε, ε, θα δεχτείτε μία μπλε κάρτα από τον συναδελφό μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, θέλω να θέσω το ερώτημα το εξής. Γιατί οι πράσινοι δεν υποστηρίζουν να ονοματίσουμε αυτή την νομοθεσία Μαγνίτσκι, νομοθεσία Μαγνίτσκι. Όχι μόνο για συμβολικούς λόγους, το είναι προφανές, αλλά επειδή είναι ένας τρόπος να ορίσουμε γιατί υπάρχει αυτή η νομοθεσία, γιατί τη χρειαζόμαστε, να στείλουμε ένα μήνυμα προς όσους χρησιμοποιούν το έγκλημα για να μπορέσουν να πλουτίσουν εις βάρος του λαού τους. Ε, γιατί λοιπόν δεν υποστηρίζεται αυτή η νομοθεσία να έχει αυτό το όνομα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και εμείς ε, στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητήσαμε διεξοδικά για το θέμα αυτό με όλες τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση ανά τον κόσμο. Έχουμε νομοθεσία ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που φέρουν αυτό το όνομα Μαγνίτσκι. Όλες οι άλλες νομοθετικές πράξεις που είναι όμως εξίσου καλές όπως στον Καναδά, όλες αυτές οι πράξεις ε, δεν φέρουν ονόματα. Θεωρώ ότι έχετε λάθος αγαπητέ συνάδελφοι όταν ισχυρίζεστε ότι η νομοθεσία αυτή δεν θα είναι εξουσιαστική αν δεν φέρει το όνομα Μαγνίτσκι. Και λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι ε, στην ε, συνεδρίαση δεν αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά στη νομοθεσία Μαγνίτσκι, όπου να γίνεται ειδική αναφορά για την επιβολή κυρώσεων. κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως και είναι κρίσιμο να ε, καταδικάσουμε ε, τις, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν είναι δουλειά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει κυρώσεις. Διότι τελικά τιμωρείτε χώρες που δεν συμφωνούν με την πολιτική σας είτε στο, ε, στο μεταναστευτικό, είτε στα θέματα των δύο φίλων, όπω στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Θέλετε ουσιαστικά να καταρρύψετε του πολιτικού σα αντιπάλου. Και αυτό είναι καταδικαστέο. Διότι τελικά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το χρησιμοποιείται για, για πολιτικούς, χαμηλά πολιτικούς λόγους και βεβαίω αυξάνονται οι πιέσει για του Ευρωπα... για και... και οι απειλέ, όπω ο Ισλαμισμό, ο ακραίο εδώ και 20 χρόνια είναι εκατοντάδε τα, τα θύματα του Ισλαμισμού στη Γαλλία. Αυτό είναι που, που απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ λοιπόν να, σκεφ, να μην αναφερθούμε στην, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, που προστατεύει τελικά του τρομοκράτε αντί να προστατεύει τα δικαιώματα. Πρόσφατα μάλιστα δεν ε, δέχτηκε να εκδιωχθεί ο Καμέλ Νταουντή, ο οποίο έχει χάσει την καλλική τυπικότητα και που αυτή τη στιγμή μένει στο ΡΙΑΚ στα έξοδα του Με έξοδα του κράτου. Επίση, απαγορεύεται η, ε, το να, μπορούμε να ψάξουμε σωματικά τους επισκέπτες στα, στις φυλακές με το πρόσφατο ατύχημα που είχαμε στη, σε μια φυλακή στη Γαλλία. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και είναι επικίνδυνο για τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Η κυρία ενα για ένα λεπτό. Όλοι γνωρίζουμε τα πλαίσια αυτού του προσχεθείου η Εστονία, η Λιθουανία, η Λετονία, ε, Καναδάς, ΗΠΑ έχουν τον αντίστοιχο νόμο τύπου Μαγνίτσκι και διώκονται ε, όσοι διαπράττουν τέτοια εγκλήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρξει μία αντίστοιχη ευρωπαϊκή πράξη και θα πρέπει να γίνει χωρίς ε, πλέον ε, αναβολές θα ήθελα η κυρία Μογκερίνη να προβάλλει μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου τύπου Μαγνίτσκι πριν από το τέλος της θητείας. Είχαμε πολλά θέματα ερμηνείας και εφαρμογής και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πρακτική. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ασής για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από αποτελεί σημείο αναφοράς σε σχέση με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου δεν υπάρχει τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως στην Ευρώπη. Η κοινωνία των πολιτών επαγρυπνεί εκεί που χρειάζεται. Όμως αυτή η αρχή θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσα που να μην αφήνει ατιμόρυτους τους ε, διαπράκτες. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό το πλαίσιο δεν είναι αποδοτικό και διεξοδικό. Χρειάζεται επιτάχυνση της διαδικασίας κυρώσεων που να είναι στόχοθετημένες, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Ο κύριος Γιούρεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι βουλευτές, η πολιτική μας θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες αρχές που είναι πολύ απλές θα πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους που είναι υπέρ των αξιών μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, οι χριστιανοί διώκονται παντού, ιδιαίτερα στην Αφρική. Γι' αυτό θα πρέπει να τηρούνται όλα τα δικαιώματα και να μην υποδαβλίζουμε πολιτικές διενέξεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να παρέμβει ως προς το ανθρωπιστικό δίκαιο, εκεί όπου υπάρχουν αδικίες, διότι εδώ δεν πρόκειται για μια καθολικότητα αρχών. Υπάρχουν άνθρωποι Πίσω από όλα αυτά υπάρχει το θέμα της Αλγερίας. Αύριο μπορεί να είναι αποφασιστικό το θέμα. Κυρία Σαργεντίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, την προηγούμενη ζωή μου και σε αυτήν όμως ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 18 χρόνια ασχολούμαι με κυρώσεις κατά της κυβέρνησης της Ζιμπάμπουε. Ήταν οι περίφημες ευφυείς κυρώσεις όμως εδώ και 11 χρόνια οι αγώνες στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη πλέον ε, δεν συνεχίζονται και ακούγοντας εδώ τους συναδέλφους καταλήγω στο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προβλέψουμε ένα νέο νέο σύστημα επιβολής κυρώσεων όπου θα προβλέπονται ειδικέ κυρώσεις για κάθε χώρα και τα πράγματα θα πλουστευτούν. Αυτά λέγονται. Δεν είναι όμως έτσι απλά. Αν δούμε ότι η Ολλανδική κυβέρνηση ναι μεν ανέλαβε κάποια πρωτοβουλία αλλά δυστυχώς δεν έχει την υποστήριξη των κρατών μελών. Η Ολλανδική κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να συνενώσει τα κράτη-μέλη, τότε διαπιστώνουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Βεβαίως μπορεί να πει κανεί ότι είναι απλά και δίνοντας ένα όνομα υποτίθεται ότι η κατάσταση διευκολύνεται, αλλά αυτό απέχει, πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Η κυρία Αρνοτού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να είμαστε υποκριτές ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πράξη Μαγνίσκη ήθελε μόνο να προβεί σε χρηματικές κυρώσεις κατά του ρωσικού καθεστώτος και ε, να μην υπάρχει παρεμβατισμός όπως ήθελαν η ειπα κάτι το οποίο δεν επιθυμούσε η Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να ε, προβάλλετε κυρώσεις λέτε, μα αυτό που θέλετε είναι να επηρεάσετε την κατάσταση αλλά αυτό πολύ υπολοιματικά θα μπορούσα να πω, αρκετή υποκρισία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη που χάνουμε και που κερδίζουμε, διότι μόνο τα κέρδη είναι ύψης της σημασίας. Έτσι κυβερνεί, κυβερνάται ο κόσμος και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μανιχαϊστική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αλαφράνκα για ένα λεπτό. από το 90, από τότε δηλαδή που μπήκε και η Αργεντινή στην ε, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια ειδική ρήτρα, ε, προβλήθηκε αυτό το ζήτημα το οποίο είναι στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δηλαδή προσδίδουμε μεγάλη σημασία στις θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η εφαρμογή που δεν είναι άμεση και η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Ε, ε, τη στιγμή που υπάρχει ο κανόνας της ομοφωνίας, όπως είπε ο Επίτροπος, υπάρχουν άλλοι που εν, μία νυχτή λαμβάνουν αποφάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας ευέλικτος ε, κατάλογος και ε, συγκεκριμένες κυρώσεις ε, τάχιστα. Αυτό είπε και η κυρία Κάνιέτε. Θα πρέπει δηλαδή να μας ε, σέβονται πολύ περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή από ό,τι ισχύει τώρα. Η κυρία Πύρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι βλέπω η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι και η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδεικνύει πάντα ότι είμαστε ενωμένοι κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται, έχουμε να κάνουμε με κατάφορη και κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πολλές φορές ε, παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Καλό είναι αυτό, είναι αποτελεσματικό. Υπάρχουν δύο μεγάλα ε, πλεονεκτήματα από τέτοιου είδους δράσεις. Αφενός προστατεύονται οι πολίτες και αφετέρου οι δράστες θίγονται στην αχύλιο πτέρνα τους. Οι κοινέ κυρώσεις εντάσσονται σε μια διαδικασία και με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται πιο ισχυρή. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι καλύτερη να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυρία Χάουταλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια υφέρπουσα κατάσταση. Έχουμε αυταρχικές ε, κυβερνήσεις. Ε, πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτές τις αλλαγές, κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρεμπιπτόντως, άκουσα τι συζητήσει που γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα και καταλήγω στο ότι στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην Ικαράγουα, στο Καζακστάν έχουμε καθεστώτα αντιδημοκρατικά και καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα δηλαδή η εργαλειοθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Άνωσης πρέπει να προσαρμοστεί. Έχουμε δράσεις, οι κυρώσεις ε, οι κατά των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για να στεφτούν από επιτυχία είναι απολύτως απαραίτητο το νέο καθεστώς να είναι υγιές και να τηρούνται υψηλές προδιαγραφές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωστή ενημέρωση. Επίσης, χρειαζόμαστε ε, το να υπάρχει και μια συνέπεια γιατί αλλιώ δεν μπορούν να υπάρξουν εγγύησει. Θέλω να σα πω ότι δεν θέλουμε να υπάρχει συμμετρία με το καθεστώ κυρώσεων ε, των ΗΠΑ, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ε, απαραίτητα δικαστικά εχέγγυα και γι' αυτό λοιπόν είμαι ευγνώμων στην ύπατη εκπρόσωπο και στο Συμβούλιο που προέβησαν σε μια ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά αυτό το νέο εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Toolbox. Είναι ένα νέο σύστημα το οποίο πρέπει να τεθεί σε και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να αποτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριο ήλστρα. Όχι, δεν είναι εδώ. Ο Κέλλα μου, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί επιτέλους αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα καθεστώς, ε, ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει να γίνει μια κοινή προσπάθεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, η πρέπει να είναι συνεπή από όλα τα κράτη-μέλη. Εμεί καλωσορίζουμε ε, το γεγονό ότι ενισχύει το κανόνα τη ομοφωνία για το θέμα αυτό. Όμω, αυτό πρέπει να γίνει υπό την προπόθεση ότι πρέπει να οδηγήσει σε επιλεκτική εφαρμογή ε, απέναντι με αυτού με του οποίου δεν συμφωνούμε. Πρέπει να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή για όλου. Για την ώρα, η πρόοδο από την απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα κατάλογο για μια νομοθεσία Μαγνέτσκι στη δεκαετία του 1990 ήταν πάρα πολύ αργή. Είχαμε το ψήφισμα του Κογκρέσου των Πολιτειών και νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να διατηρήσει το όνομα Μαγνίτσκι ε, που έχει μια συμβολική καθολική αξία. Επίσης είναι ντροπή το γεγονός ότι η Ρωσία ως τώρα δεν περιλαμβάνεται ε, την μαύρη λίστα για το ξέφλυμα μαύρου χρήματο και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ανδρουλάκη έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Παραμένει η κύρια δύναμη υπεράσπιση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συζήτηση για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε ανθρώπου ή κυβερνήσει παγκοσμίω που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια μεγάλη πρόκληση και πρέπει όλοι σήμερα να απαντήσουμε θετικά για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας ανάμεσα στους λαούς που επιζητούν την ευρώπη της αλληλεγγύης της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. για να είναι όμως αποτελεσματικό θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην λειτουργεί με την αρχή της ομοφωνίας. δεν μπορούμε να είμαστε έρμεοι πολιτικών και εθνικών συμφερόντων όπως συμβαίνει πολλές φορές στο κοινοβούλιο όσο και στο συμβούλιο. το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα και κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς κάνουν ότι δεν βλέπουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες της μέσης ανατολής όπως από την άλλη πλευρά η ευρωπαϊκή αριστερά δεν πιστεύει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή και ανθρωπιστική κρίση στην βενεζουέλα των τριών εκατομμυρίων προσφύγων και της έλλειψης βασικών αγαθών. τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως δεν είναι πεδίο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. η υπεράσπιση τους πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο προβάλλει ένα σφαιρικό καθεστώς ε, κυρώσεων. Όπως ε, έκαναν η ΙΠΑ, ο Καναδάς και όλες οι βαλτικές χώρες. Μία νομοθετική πράξη τύπου Μαγνίτσκι ε, άρα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΙΕΔ να προετοιμάσουν μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για μία πράξη τύπου Μαγνίτσκι για να γίνει πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και να μην επιτρέπεται η είσοδος σε τέτοιους πολίτες του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προβάλλουμε ένα κυρωτικό καθεστώς όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Διαφορετικά θα ε, μειωθεί η ηγετική μας θέση. Ε, Ροντρίγκες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν μπορεί να υπάρχει ατιμορρησία για αυτούς οι οποίοι καταδικάζουν άλλους λόγω έλλειψης ανέξη Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δολοφονία δημοσιογράφων ή εξόντωση ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δίνει καταφύγιο σε περιπτώσεις τέτοιων παραβιάσεων. Θα πρέπει να έχουμε μία νομοθετική πράξη που να αποτρέπει την είσοδο αυτών που παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να τους χορηγούμε θεωρήσεις. Δεν μπορεί να τους δεχόμαστε στο σπίτι μας. Χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη πρόταση μεγάλης εμβέλειας εάν δεν θέλουμε να έχουμε ε, ένα γράμμα κενό περιεχομένου. Δεν μπορούμε να ε, σπηλώσουμε την μνήμη αυτών που χάθηκαν. Κάτσετε άι τώρα. Έχουμε επτά συναδέλφους. Θα λάβετε το λόγο όλοι, αλλά θα ήθελα να αρκεστείτε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Ντρογεύσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν πιστεύω στις κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι είναι και η μόνη λύση, το μόνο μέσο ή εργαλείο για να ασκήσουμε πίεση, ούτε πιστεύω στη δύναμη των ψηφισμάτων. Έχουμε ένα πληθωρισμό ψηφισμάτων που δεν είναι αποδοτικά. Εγώ είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας με τη Λευκορωσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, αλλά να προβάλλουμε και έναν διάλογο, να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών. Είμαι κατά του πληθωρισμού ψηφισμάτων για κυρώσεις που σχετίζονται με άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε έτσι να φτάσουμε σε αποδοτικό αποτέλεσμα. κύριος Μαυρίδης. Είστε Μαυρίδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θέλω και εγώ με τη σειρά μου να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό επιβολής κυρώσεων ο οποίος να στοχεύει και σε άτομα εγκληματίες όσο και σε κυβερνήσεις κρατών. το ζητούμενο όμως είναι ο μηχανισμός αυτός να είναι αποτελεσματικός και αμερόληπτος. είτε τα εγκλήματα διαπράττονται εντός ευρωπαϊκής ένωσης είτε εκτός ευρωπαϊκής ένωσης είτε ο παραβάτης είναι στη ρωσία είτε είναι στην τουρκία. δυστυχώς η συμπεριφορά μας μέχρι σήμερα θα δείξει στην πορεία αν θα αλλάξει και θα αντιμετωπίσουμε επιτέλους όλους αυτούς τους παραβάτες με τον ίδιο τρόπο. πάντως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχει φανεί έχει καταφανεί ότι δεν αντιμετωπίζουν τους παραβάτες και εγκληματίες με τον ίδιο τρόπο. για παράδειγμα και τελειώνω το έγκλημα της εξαφάνισης του χριστιανικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού στο βόρειο τουρκοκατεχόμενο μέρος της κύπρου είναι έγκλημα για το οποίο σιωπάτε κύριε επίτροπε. Κυρία Τόμασιτς, για ένα λεπτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται από πολλές τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές σχέσεις. Οι ευρωπαϊκοί ηγέτες μιλάνε για μια κοινότητα αξιών, αξιών που διέπουν όλη μας την πορεία, αλλά αυτό δεν ισχύει έμπρακτα, γιατί υπάρχουν παραβιάσεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό υπάρχει και το ΕΔΑΔ και δεν χρειαζόμαστε άλλο μηχανισμό. Υπάρχει αυτός ο κυρωτικός μηχανισμός εκείνων που δεν διέπονται από το όραμα των Βρυξελών. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι φεντεραλιστές. Θα πρέπει να έχουμε αποδοτικούς μηχανισμούς προς τρίτες χώρες. Ο κύριος Σολέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για να μπορέσει να είναι αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν λέτε προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο, δεν φτάνουν τα λόγια. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα όργανα, εργαλεία. Αυτό το καθεστώ κυρώσεων προ άτομα ε, από κρατικού και μη κρατικού φορεί ε, που είναι υπεύθυνοι για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητο. Είμαστε στην πρώτη γραμμή ε, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι αυξάνεται η ορατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω ένα υπεύθυνο διεθνή παράγοντα. Στέλνουμε ένα χειρό μήνυμα προ τι δικτατορίε, ε, στα αυταρχικά καθεστώτα που υπάρχουν ακόμα και που συστηματικά παραβλέπουν τα δικαιώματα και το καθήκον να προστατεύσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει να δυσκολέψουν λίγο περισσότερο τη ζωή αυτών ε, που είναι υπεύθυνοι για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι καταχρήσει πρέπει να υποστηρίξουμε τα θύματα αυτών των καταχρήσεων, αλλά και αυτού που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Για όλου του λόγου, ε, ζητώ από το Συμβούλιο να φτάσει σε συμφωνία για αυτήν, αυτό το καθεστώ το οποίο είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ο κ. Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Συνάδελφοι, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κάποιου είδους κυρώσεις οι κυρώσει όμω αυτέ πρέπει να υλοποιούνται μετά από μια ενδελεχή και δημοκρατική συζήτηση με το κράτο κατά του οποίου επιβάλλονται. σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην πείσουμε το υποσυζήτηση κράτο ή του αξιωματούχου του αλλά χωρίς αμφιβολία θα έχουμε καταφέρει να αναπτυχθεί η αναγκαία συζήτηση μέσα στον πληθυσμό αυτού του κράτου. χωρί αυτή τη δημόσια συζήτηση μπορεί εύκολα οι κυρώσει να εκλαμβάνονται από αυτό το κράτο ω εχθρική κίνηση και αυτό δεν θα είναι καθόλου επικοδομητικό. ευχαριστώ. Σήμερα η παγκόσμια τάση οδηγεί στο να υπονομεύεται το διεθνέ δίκαιο, κυρίω όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολυμέρεια δέχεται επιθέσει από μία σειρά κρατών, οι προηγούνται και είναι επικεφαλή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι λοιπόν σημαντικό η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ε, το καθεστώ αυτό το ευρωπαϊκό των κυρώσεων ε, προχωράει οι κυρώσει μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι όμω απαραίτητο οι κυρώσει να είναι στοχευμένε, να υπάρχει συνέπεια και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Πρόοδο λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μου υπενθυμίζει ότι αν υπάρξει Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορέσει να συμμετέχει σε αυτέ τι ε, θετικέ πολιτικέ. Από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει για το Brexit, η συντηρητική κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία δείχνει κινησμό, όλο και περισσότερο περισσότερο κινησμό. Η κυρία Μέη, ε, συμμαχία με τον Τραμπ και τον Ορμπάν. Σήμερα Βλέπουμε ότι υπάρχει και συνεργασία με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων. Ε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία των 27 κρατών και αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να έχουμε ένα απομονωμένο, απελπισμένο νησί. Κυρία Μιράντα, κυρία Πρόεδρε, ένα σύστημα ακυρώσεων ε, ε, εμείς είμαστε υπέρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαραίτητο. Αλλά ε, ταυτόχρονα δεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση όπου είμαστε συνένοχοι απέναντι στην ατιμορρυσία. Θα δώσω τρία παραδείγματα. Μαρόκο, την περίπτωση του ΡΙΦ, μόλις πρόσφατα Χθε καταδικάστηκαν διάφοροι ακτιβιστέ στο ΡΙΦ που είχαν υποθεσπιστεί κοινωνικά δικαιώματα, ελευθερία έκφραση. Να σα δώσω και άλλα παραδείγματα, κύριε Επίτροπε. Η περίπτωση τη Δυτική Σαχάρα όπου υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι κάνουν απεργία πείνα. Και βεβαίω η περίπτωση τη Τουρκία. Θα μιλήσουμε αργότερα για την Τουρκία βέβαια, αλλά υπάρχουν πολιτικοί ηγέτε που είναι στη φυλακή, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι. Και τι να πούμε για το Ισραήλ, κύριε Επίτροπε, τι να πούμε για το Ισραήλ. Θα θέλαμε λοιπόν να, σταματήσει αυτή η συνενοχή, ε, διότι και οι εμπορικέ ε, συμφωνίε που κάνουμε παράδειγμα με τι χώρε αυτέ ε, είναι επιβλαβεί αυτά που συνέβησαν με την, την μεγάλη ε, πορεία για την επιστροφή των Παλαιστινίων στο, στα κατεχόμενα εδάφη ε, είναι εγκλήματα και 35 εκ των θυμάτων είναι παιδιά και εκατοντάδες είναι νεκροί. Τι θα κάνουμε για αυτά λοιπόν. Θα ήθελα ο Επίτροπος, ο κύριος Σαχάν, να λάβει το λόγο για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να πω ένα θερμό ευχαριστώ ε, σε αυτή την ε, ιδιαίτερα χρήσιμη και επίκαιρη ανταλλαγή απόψεων και δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω και πάλι για όλες τις παρεμβάσεις, για τα σχόλιά σας, για τις προτάσεις σας. Η σημερινή συζήτηση για άλλη μια φορά καταδεικνύει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ένα οικουμενικό ε, σύστημα επιβολής κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίω πρέπει να υπάρξουν και περαιτέρω μελέτε. Όπω ε, αναφέρθηκε, οι συζητήσει ε, εστιάζουν στα ανοιχτά θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε βάθο για να έχουμε μια τεκμηριωμένη πολιτική άποψη κατά πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα. Οι συζητήσει θα συνεχιστούν στο Συμβούλιο. Ε, θα συνεχίσουμε επικοδομητικά να καταλήξουμε κάπου ομόφωνα. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημασία που αποδώσετε σε αυτό το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. με τον ε, πίτροπο. Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος με βάση τις δηλώσει που έχουν γίνει. Κλείνει αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη. Περνάμε στο επόμενο θέμα, την έκθεση της κυρίας Πύρη σε σχέση με την κατάσταση στην Τουρκία. Έκθεση του 2018. Περιμένουμε την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Τσόκ, η οποία θα έρθει τα επόμενα λεπτά και δίνω το λόγο στην κυρία Κάτι Πύρη για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να βρίσκεται κανείς ε, για 17 μήνες στη φυλακή χωρίς να ξέρει τι πράγμα κατηγορείται, αυτή είναι η πραγματικότητα στη σημερινή ε, Τουρκία. Τον Οκτώβρη του 2017 συνελήφθη ο λόγο λόγω κατηγορούμενος ε, ένας, μια εμβληματική προσωπικότητα της τουρκικής κοινωνίας, άσκησε κριτική κατά του Ερντογάν, ε, ο ΣΜΑΝ και άλλοι κρίνονται κατηγορούμενοι για το ότι θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση ε, και αντιμετωπίζουν την ποινή της κάθριξης, ε, διαβίου κάθριξης. Απλά αυτοί συμμετείχαν σε μία διαδήλωση αυτό κρίθηκε ότι ήταν μια διεθνή σκευωρία για να ανατραπεί η κυβέρνηση. Τα στοιχεία κατά του Οσμάν Καβαλά ήταν από κάποια ε, υποκλαπέντα τηλεφωνήματα όπου ε, αναφέρει ότι θέλει να ε, μετατρέψει κάποια προϊόντα, αλλά αυτό που δεν είναι δεν αρκεί. Ε, θα μπορούσε κανείς να γελάσει για όλα αυτά αν τα πράγματα δεν ήταν σοβαρά. Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο έχει κατρακυλήσει η δημοκρατία στην Τουρκία. Τώρα λοιπόν, ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά. Ποια είναι η απάντηση στην κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη γειτονική χώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προηγείται όχι μόνο στο να τοποθετείται, αλλά ζητώντα και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο να εκμεταλλευτούν ό,τι έχουν στη διάθεσή τους για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στον κύριο Ερντογάν να μην υπάρξει περαιτέρω διολίστηση και από την άλλη να δείξουν στους Τούρκους πολίτες ότι είμαστε θεματοφύλακες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι είμαστε στο πλευρό τους. Μέχρι τώρα όμω οι Ευρωπαίοι ηγέτη δυστυχώ δεν τα έπραξαν αυτά που έπρεπε να πράξουν. Η Τουρκία έχει εξαφανιστεί από την προσοχή μα, δεν βρίσκεται πια στι ειδήσει παρά μόνο όταν πρόκειται για πολίτε τη Ένωση. Φαίνεται ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν αποδεχτεί την κατάσταση στην Τουρκία, ε, οι δικέ μα εκκλήσει για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο προσκρούν σε ότα μία κόντων στην Τουρκία, αλλά και σε ε, Μητροπόλεις ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έχουμε ξεπεράσει όλες τις κόκκινες γραμμές. Συνεχίζεται η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Η Τουρκία φυλακίζει δημοσιογράφους και πάνω απ' όλα το νέο σύνταγμα σταθεροποιεί το αυταρχικό καθεστώς του Ερντογάν. Για το λόγο αυτό ζητάμε από το Συμβούλιο επίσημα να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας. Δεν θα μπορούσε προφανώς να υπάρξει ένταξη ως έχουν σήμερα τα πράγματα, αλλά το να συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ένταξη μεταξύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχίζουμε τον πρόεδρο Εντρογάν, αυτό είναι παροδία. Ε, θέλουμε να μα πει τι θα κάνει για τον Οσμάν Καβαλά ή για τον Ντερμιτάς ε, ή για τον αρχηγό τη αντιπολίτευση που ήταν στη φυλακή για δυόμιση χρόνια και για άλλα μέλη του Κοινοβουλίου και μέλη των ΜΚΟ για δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων που καταδικάστηκαν χωρί ε, δίκαιη δίκη για του ακτιβιστέ ε, των ΛΟΑΔ, για πολλού που δεν έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, για τις στην Τουρκία που στην ημέρα της γυναίκας βγήκαν στους δρόμους και είχαν να αντιμετωπίσουν τις πλαστικές σφαίρες της αστυνομία. Η σιωπή του Συμβουλίου δίνει νερό στο μήλο του Ερντογάν. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να καταλήξουμε με μια στρατηγική. Αυτή την Παρασκευή μπορεί να ξεκινήσει αυτό όταν θα υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Και κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μετά από αυτά τα πέντε χρόνια να ευχαριστήσω ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους σκιώδεις συζητητέ που συνεργάστηκαν μαζί μου για το θέμα αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια. Πολύ καλή αγαστή συνεργασία και θέλω να ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να ενώσουμε το Κοινοβούλιο να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους Ευρωπαίου ηγέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα η κυρία Τσότ να λάβει το λόγο εξ του Συμβουλίου. το μικρόφωνο σας. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πολύ στην πρόσκληση για τη σημερινή συζήτηση να συζητήσουμε ε, την έκθεση του 2018 για την Τουρκία και να δούμε θέματα αμοιβαίας ε, μέρημνας και ανησυχίες. Λαμβάνουμε υπόψη τα σαφή μηνύματα που ανακύπτουν από το ψήφισμά Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Τουρκία, ιδιαίτερα την ε, αναθεώρηση του συντάγματος που μας ανησυχεί γιατί όπως ε, είδατε ήδη υπάρχει αυτή η ολίσθηση σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη ρίση θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων όπως ε, είδαμε και στην έκθεση του 2018 σε σχέση με τη μελλοντική πορεία της διεύρυνσης. Αυτό το είδαμε και πέρσι καθώς και με τη σημερινή έκθεση του Κοινοβουλίου στις 18 Ιουλίου 16 το Συμβούλιο καταδίκασε το πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016 και τάχθηκε υπέρ των δημοκρατικών αρχών. Βεβαίως η Τουρκία Τουρκία αντιμετώπισε μία απειλή, αλλά είναι δυσανάλογα τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν μετά από την απόπειρα πραξικοπήματος, κάτι το οποίο δυστυχώς μας οδηγεί στο να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Η Τουρκία απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή της πορεία πλέον. Ε, ε, δέχομαι το αίτημά σας για την αναστολή διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, αλλά το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Ιουνίου 18 θεώρησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση φτάσανε σε αδιέξοδο για τους λόγους που προαναφέρατε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κλείσουμε την πόρτα στην Τουρκία, να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθήσουμε έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία, διότι είναι βασικός μας εταίρος σε πολλούς τομείς και αυτό είναι προς αμοιβαίο συμφέρον. Αναφέρομαι στις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε και την ανάγκη συνεργασίας κοινού συμφέροντος και ενδιαφέροντος όπως τη μετανάστευση, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ενέργεια, εμπόριο και ούτω καθεξής. Η διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Η κοινή αυτή διαχείριση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τάσεται υπέρ και των δύο μερών, όπως ορίστηκε ήδη από το 17. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πολλούς μετανάστες που προέρχονται από την Τουρκία, παράνομους μετανάστες και βεβαίως υπάρχει και η προσφυγική ροή των Σύρων. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Τουρκία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και συνεργάζεται επικοδομητικά η χώρα αυτή. Παράλληλα, η Τουρκία θα πρέπει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Κύπρο με βάση το επιπρόσθετο πρωτόκολλο στην ε, Συμφωνία Σύνδεσης. Εμείς ως Προεδρία θα συνεχίσουμε να θίγουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα με τους συνομιλητές μας από την Τουρκία σε κάθε επίπεδο και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πείσουμε την Τουρκία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό Τσότ και θα ήθελα τώρα ο Επίτροπος Χάν να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια Κάτι πύρη, αλλά και όλους τους σκιώδεις όλων αυτών των ετών για την εξαιρετική σας εργασία υπέρ αυτής της υποψήφιας για προσχώρηση χώρας. Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε αναγνωρίσει πολλά δεινά στην ετήσια έκθεση για το 18 και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την τάση της ε, ε ηγεσίας της Τουρκίας. Η δίωξη του Οσμάν Καβάλα και πολλών άλλων δημοσιογράφων δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ως προς την προστασία της κοινωνίας των ε, πολιτών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο δεν υποστηρίζεται στην Τουρκία. Η Τουρκία ε, θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στην Τουρκία και στυλιτεύουμε την όλη κατάσταση όταν παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γιατί η Τουρκία θα πρέπει να προβεί στις δέουσες μεταρρυθμίσεις. Όμως η Τουρκία είναι εταίρος και γειτονική χώρα και συνεργαζόμαστε σε τομείς όπως η ενέργεια, καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, εμπόριο και αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό ανά τον κόσμο και βλέπουμε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ μας. Επίσης, πρόσφατα υπήρξαν ε, πολλές ε, αλλαγές και θετικά ζητήματα ως προς τον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου και θα γίνει φυσικά και μια νέα συνάντηση όπως προβλέπετε αργότερα αυτή τη βδομάδα. Στις 22 Νοεμβρίου στην Άγκυρα η ύπατη εκπρόσωπος και ο υποφαινόμενος τονίσαμε στην Τουρκία ότι θα πρέπει να αλλάξει στάση εάν θέλει πραγματικά να βελτιωθούν οι σχέσεις μας. Κατά τον πρόσφατο διάλογο ε, αξιωματούχων για οικονομικά ζητήματα, ο αντιπρόεδρος ε, Κατάινεν στηλίτευσε την δίωξη δημοσιογράφων. Η Τουρκία θα πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις με όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα με την Κύπρο. Τονίσαμε το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να προβαίνει σε προκλητικές δράσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Θα πρέπει να τίνουμε χείρα βοηθείας προς αυτούς τους διοκόμενους ε, πληθυσμούς. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζόμερ έχει τώρα το λόγο για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κάτριν Πούρη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω και του σκιώδη ηγητέ των άλλων πολιτικών ομάδων. Τελικά καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο, το οποίο χρήζει μόνο κάποιων μικρών βελτιώσεων σε ένα σημείο συγκεκριμένα, στο σημείο εκείνο, όπου αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσει πρέπει να ανασταλούν. Αυτό το αίτημα δεν είναι καινούργιο καινούριο. Εμείς ε, το γνωρίζαμε, το είχαμε φυλάξει για την περίπτωση εκείνη όπου θα καταργηθεί η δημοκρατία στην Τουρκία. Όμω με τον τρόπο αυτό δεν εντυπωσιάσαμε την Τουρκία. Ε, το Σύνταγμα τροποποιήθηκε, καταργήθηκε το κράτο δικαίου και ακόμα και αν ανασταλούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ε, παρόλα αυτά η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει δικαίωμα για τα κονδύλια τα προενταξιακά. Με αυτά τα χρήματα όμως κατ' ουσίαν στηρίζουμε την κυβέρνηση τη Τουρκία. Τουρκία, η οποία καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, διώκει του αντιπάλου μέχρι και στο εξωτερικό, επιβάλλει υψηλέ ε, ε, κυρώσει, ε, κυνήγι μαγισσών κατά των οπαδών του Γκυλέν τα επιθυμούμε όλα αυτά. Η δική μου πολιτική ομάδα λέει ότι πρέπει πλέον να σταματήσουν διαπαντός οι διαπραγματεύσεις και στην περίπτωση αυτή τα προεντιεξιακά κονδύλια μπορούμε να τα διοχετεύσουμε στην κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επουδενή δεν μπορεί να δεχτεί και άλλη διεύρυνση. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να μας στηρίξετε στο κείμενο και να ζητήσουμε την πλήρη πλήρη πάυση, την διακοπή και όχι μόνο την αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την Προεδρία τη Ρουμανία για την πολύ ισορροπημένη αξιολόγηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία διεύρυνση μα έχει επιτρέψει να επηρεάσουμε σημαντικά ε, τον δρόμο τη Τουρκία προ τη δημοκρατία τι τελευταίε